προϊόντα διτής, διπλής χρήσης. Και τώρα θα λάβει τον λόγο ο ίδιος ο εισηγητής. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Φιέρνερ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν θα εξαντλήσω το σύνολο του χρόνου των τεσσάρων λεπτών. Κατά το τέλος της συζήτησης θα ήθελα να μπορέσω κάποια ερωτήματα να απαντήσω αν χρειαστεί από πλευράς χρόνου. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι αυτή η έκθεση έχει τον εξή στόχο. Θέλουμε με αυτήν οι νόμοι μας, οι διατάξεις και οι ρυθμίσεις να προσαρμοστούν στις αλλαγές, στις μεταβολές που απέρευσαν λόγω της νέας συνθήκης. Εδώ πρόκειται λοιπόν για ένα κάπως περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα θέμα. Πρέπει μια επιτάχυνση να μπορέσει να διασφαλιστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα κατανόησε ότι κατ' εντολή τέτοιες εξουσιοδοτήσεις ε, για ε, εκτέλεση τέτοιων πράξεων απαιτείται για να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο δεν θα αντιμετωπίζει μεγάλους καταλόγους που θα απαριθμούν ατέλειωτα τέτοια προϊόντα και τα οποία θα πρέπει όλα να ελέγχει κατά περίπτωση. Αυτό που θέλουμε είναι είναι αυτές οι μεταβολές να μπορέσουν με σύντομο, γοργό τρόπο να αντιμετωπίζονται και να διευθετούνται, διότι διαφορετικά οι κατάλογοι, οι πίνακες αυτοί δεν θα είναι επίκαιροι και δεν θα έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Για τις αλλαγές μέχρι το 2010 αναφερόμαστε, δηλαδή πρέπει ταχύτατα να μπορούμε να αντιδράσουμε, ώστε όλες οι αλλαγές που από το 2011 ε, έχουν απορρεύσει ενδιάμεσα να μπορέσουν και αυτές να καλυφθούν και να διευθετηθούν. Έχουμε ωστόσο μια ολόκληρη σειρά δυσχεριών που πρέπει να υπερβούμε, να ξεπεράσουμε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή. Πάρα πολλές απόψεις αφορούσαν όχι μόνο τα τεχνικά θέματα και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά πιστεύω ότι εμείς οι ίδιοι μια ολόκληρη σειρά άλλων θεμάτων και ζητημάτων αντιμετωπίσαμε και από πλευράς των σοσιαδημοκρατών, των σοσιαλιστών το κατανόησα με τέτοιο τρόπο ότι διαφορετικές προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν για θέματα διαφάνειας ε, της ε, διασφάλισης ε, των συγκεκριμένων πτυχών κτλ. Έχουν τη σημασία τους αυτά τα θέματα, αλλά δεν θέλω να διακυβεύσουμε με αυτό το έγγραφο να καθυστερήσουμε και να παραταθεί η συνολική αυτή διεργασία. Θέλουμε οι, εμείς οι σοσιαλιστές να επιταχυνθούν τα πράγματα, διότι το συνολικό, ο συνολικός κατάλογος προϊόντων διαρκώς μεταβάλλεται και είναι σημαντικό να υποβληθεί μια πρόταση από την Επιτροπή σε σχέση με το 2013 για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ουσιαστικά δεν βλέπω να υπάρχουν λόγοι για τις τροπολογίες ε, που θέλει να εγκριθούν η σοσιαλιστική ομάδα. Είναι περισσότερο περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα θέματα αυτά. Ιστερότερα, μεταγενέστερα μπορούμε να καταλήξουμε σε μια σειρά προσαρμογών και να καταλήξουμε σε αυτές τις ρυθμίσεις που επιθυμούν οι σοσιαλιστικοί συνάδελφοι. Αυτό αφορά το περιεχόμενο τη εκθεσή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεχούχτ έχει τώρα το λόγο. Uh, uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Η πρόταση την οποία εξετάζουμε σήμερα αφορά την διτή χρήση ορισμένων ε, προϊόντων και φυσικά η πρόταση αυτή αφορά την ίδια μας την ασφάλεια. Έχει σαν στόχο να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αποτελεσματική στο να αποτρέψει το κίνδυνο της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής και την στρατιωτική χρήση προϊόντων για πολιτική χρήση και με τον τρόπο αυτό πρέπει να συμμορφωθούμε και με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις στον τομέα αυτό. Δεύτερον, η πρώτη στάση αυτή αφορά την, στην ευμάρειά μας. Θα δημιουργήσει ένα ισόπεδο πεδίο ανταγωνισμού σε σχέση με τους ανταγωνισμούς μας, με τους ανταγωνιστές μας και θα εξασφαλίσει ότι οι έλεγχοι εξαγωγών δεν θα θίξουν νευραλικούς τομείς της εξαγωγικής μας βιομηχανίας. είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ μια στεναρή αμυντική βιομηχανία και την προώθηση των εξαγωγικών μα συμφερόντων. Ώστε να επιτύχει του στόχου αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνεται να εκχωρηθούν στην Κομισιόν οι αρμοδιότητες με το λεγόμενο κατάλογο ελέγχου για, τις, για τα προϊόντα αυτά που έχουν διπλού διτή χρήση. Η επικαιροποίηση η επικαιροποίηση αυτού του, του καταλόγου για να συμμορφωνόμαστε με τις διεθνείς μας υποχρεώσεις θα γίνεται με έναν τρόπο αυτόματο και έτσι θα ενσωματώνονται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια θέματα τα οποία πρέπει να γίνονται με τακτικό χαρακτήρα και επομένω δεν προσφέρονται στη διαδικασία νομοθεσίας. Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να, να ε, αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον κοινό κατάλογο ελέγχου. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε εμπορικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που δεν μπορούν να συναλλαγούν σε ορισμένες αγορές ενώ οι ανταγωνιστές τους μπορούν να το κάνουν γιατί ενημερώνονται πιο τακτικά οι κατάλογοι ελέγχου σε άλλες χώρες. Προτείνεται επίσης η Κομισιόν να αναλάβει την επικαιροποίηση του παρατήματος 2 του καταλόγου μας για προϊόντα διητής χρήση που επιτρέπει να αποστέλλονται τέτοια προϊόντα σε ορισμένου προορισμού χαλού κινδύνου. Πολλές φορές όμως πρέπει να αντιμετωπίζουμε ραχδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες, εμπλέκονται θέματα ασφαλείας και επομένως το ερώτημα είναι πόσο χρόνο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιβάλλει ενισχυμένους ελέγχους εάν επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας σε μια χώρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαφές ότι είναι σημαντική η ταχεία αντίδραση και η διαδικασία αυτή εξουσιοδότηση θα επιταχύνει τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, Έχω καταγράψει τι διάφορε τροπολογίε οι οποίε κατατέθηκαν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να σα υπενθυμίσω την ε, αναθεώρηση στην οποία έχει αποδηθεί η Κομισιόν σε σχέση με το καθεστώ ελέγχου προϊόντων διτής χρήση, που είναι και το κατάλληλο πλαίσιο για να συζητήσουμε θέματα τα οποία εκφεύγουν του πλαισίου του προτινόμενου κανονισμού. Όπω ανέφερα και εξήγησα προηγουμένως, μέσω του κανονισμού αυτού θέλουμε να εισαγάγουμε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία να υπάρχει ένας κατάλογος ελέγχου για την Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτει όλα τα προϊόντα διτής χρήση που μπορούν να δώσουν δηλαδή σε στρατιωτική χρήση και προϊόντα μαζικής καταστροφής. Έτσι θα εξασφαλίσουμε την ισότητα ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς μας. Αυτό διακύβευεται και σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Κάσπαρη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα εγώ να συνεχίσω εκεί που έκλεισε ο Επίτροπος Δεχούχτ. Είναι προς το κοινό μας συμφέρον να μπορέσουμε με ένα αποτελεσματικό τρόπο να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει έλεγχος και δεν αφήνουμε προϊόντα να μπαίνουν στην... να μην υπάρχει έγκριση προϊόντων τα οποία έχουν παρουσιάζεται η χρήση τους με λαθασμένο τρόπο ή με ψευδή τρόπο και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει και ε, αμφιβολία για ορισμένα προϊόντα τα οποία είναι σαφές ότι έχουν μονάχα πολιτική χρήση όπως εξαρτήματα αυτοκινήτων, υπολογιστές κτλ. Αυτό το οποίο ακόμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το θέμα του αν θα πρέπει να είναι εξάντε ή εξπόστ η εξέταση μιας εξαγωγικής διαδικασίας και αυτό μας οδηγεί σε η πρόταση η οποία υπάρχει μας δημιουργεί αμφιβολίες γιατί λέμε ότι αν ένα προϊόν βρίσκεται στον κατάλογο στη χώρα του, τότε μπορεί μια χώρα, μπορούν οι χώρες με διαφορετικούς καταλόγους ελέγχου να βοηθήσουν τους εξαγωγείς της δικής τους χώρας να ε, εξαγάγουν τα δικά τους προϊόντα. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια εξέταση είτε εξ είτε εξάντε που δεν έχει να κάνει καθόλου με το αν ένα προϊόν εξάγεται ή όχι. Το θέμα είναι αν μπορεί να υπάρξει μια σωστή δυνατότητα ανταγωνισμού για τους εξαγωγείς μας και να μην οδηγούν οι κατάλογοι αυτοί ελέγχου σε μειονεκτήματα ανταγωνισμού για του δικού μα εξαγωγεί. Φυσικά είμαστε όλοι σύμφωνοι επί τη ουσία, θα πρέπει να έχουμε καλύτερο έλεγχο, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη και ταχύτερη δυνατότητα αντιμετώπιση αλλαγή κατάσταση και γι' αυτό όπω είπε και ο εισηγητή, είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να μπορεί η Κομισιό να αλλάζει του κανόνε τους κανόνες και τους καταλόγους ελέγχου επί τη βάση των αλλαγών που γίνονται στο διεθνές σκηνικό. Ευχαριστώ πολύ για τους σοσιαλιστές. Ο κύριος Λάιχτ Φρίντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, βλέπουμε ότι όταν πρόκειται για αυτό το θέμα της, ε, των ειδών διπλής κρίσης, ε, στο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών ανάβουν τα τηλέφωνα. Γίνονται παρεμβάσεις, ε, καταβάλλονται προσπάθειες να πιστούν οι συνάδελφοι να μην ταχθούν υπέρ ελέγχων που γίνονται πριν από τις εξαγωγές. Εφόσον λοιπόν συζητάμε για το θέμα αυτό, πρέπει να πούμε περί τίνος πρόκειται. Δεν πρόκειται για καρέκλες γραφείου, όπως είπε ο συνάδελφος, αλλά πρόκειται για όπλα, πρόκειται για επικίνδυνες χημικές ουσίες και για λογισμικά. Ε, το λογισμικό που εξάγεται από την Ευρώπη αυτό ακριβώς είναι το λογισμικό το οποίο πριν από ένα χρόνο δολοφόνησε ανθρώπους στη Μέση Ανατολή. Γιατί με τον τρόπο αυτό έγιναν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώχθηκαν οι αμήντορες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν και δυστυχώς ε, για άλλη μια φορά θα πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε για το κατά πόσο αυτές οι εξαγωγές θα πρέπει να ελέγχονται εκ των προτέρων. Για τη τελική ανάλυση τι νόημα η δημοκρατία το να γίνεται η κοινοποίηση πριν ή μετά. Δεν πρόκειται για γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά για μεγαλύτερη ασφάλεια για ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από την εξαγωγή αυτών των προϊόντων και υποφέρουν από το ότι ορισμένες εταιρείε προσπορίζονται μεγαλύτερα κέρδη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η βιομηχανία της Ευρώπης να εξάγει αντικείμενα, αλλά να προβαίνει σε καλούς ελέγχους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι σοσιαλδημοκράτες ενδιαφερόμαστε να ακολουθηθεί η κατεύθυνση που σας σκιαγράφησα. Κατανοώ την Κομισιόν και το ΕΛΚ επιθυμούν όλα να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα και χωρίς πρόβλημα, όμως τα προβλήματα που προκαλούνται είναι πολύ σημαντικότερα από τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε. Μας πιέζει ο χρόνος. Γι' αυτό περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Σάκε. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στη συζήτηση για τα προϊόντα διπλής χρήσης θα ήθελα να επικεντρωθώ στις τεχνολογίες που διαδραματίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των πολιτών και μπορούν να διαρρήξουν μονοπόλια, πληροφορίες, ε, εξουσίας ε, και δίνουν πολλές κοινωνικές ε, και πολιτιστικές αναπτυξιακές δυνατότητες. αφορούν όμως και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, Βερμανία, Συρία, στην Αφρική με τη χρήση smartphone μπορούν να ασκήσουν τα ανθρώπινα, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία έκφρασης, τους συνεταιρίζεστε πρόσβαση στις πληροφορίες και μπορεί να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όποιοι φοβούνται όμως ότι θα χάσουν τον έλεγχο, φαίνεται ότι πιέζουν ε, και, κατα... και καταπιέζουν τον κόσμο με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ακτιβιστών και δημοσιογράφων ε, που τους κατασχέθηκαν ε, τα τηλέφωνα τα... Ή, ή έχουν παραβιαστεί οι λογαριασμοί τους στους ε, υπολογιστές τους είναι θέματα ζωής και θανάτου για τους ανθρώπους αυτούς τέτοιου τους θέματα και πολύ συχνά οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για να καταπιέζουν και να καταστήλουν τον άνθρωπο έχουν δυστυχώς μια ετικέτα, το Made in Europe. Οι τεχνολογίες αυτές κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εξάγουμε τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, και να, ως boomerang και να στραφούν κατά της Ευρώπης. Θα πρέπει να σταματήσει το εμπόριο των ψηφιακών όπλων. Μεγαλύτερη λογοδοσία, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού και καλύτερη ενημέρωση ώστε να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγετικό ρόλο στον όλο και πιο συχνά και ραγδαία εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο κόσμο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Φραντσίσκα Κέλλερ για τους πρασίνους. Πολλές φορές ε, τα ε, αντικείμενα διπλής χρήσης μοιάζουν αυτό, αλλά μπορούν να είναι τόσο επικίνδυνα όσο και τα πολυβόλα όπλα και τα τεθωρακισμένα. Μόνοι μας ε, υπονομεύουμε τους στόχους μας, οποτεδήποτε στέλνουμε τέτοια όπλα, τα οποία μπορούν να καταστήλουν δημοκρατικά καθεστώτα. Τα λογισμικά της Nokia ήταν εκείνα τα οποία χρησιμοποίησαν οι Ιρανοί όταν κατέστηλαν τις ε, διαμαρτυρίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι ε, βασανίστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο. Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα από τα πολλά. Και προστίθεται και το εξή ε, η Κομισιόν με τον κατάλογο που έχει για μια ανταγωνιστική βιομηχανία προάγει αυτά τα ύποπτα αντικείμενα, τα ύποπτα προϊόντα. Ε, στόχος είναι να υπάρχει ασφάλεια ε, γιατί υπάρχει κίνδυνος ε, προς όφελος μιας αμφιλεγόμενης βιομηχανικής πολιτικής να καταστέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να τα ξεπουλάμε τα έλεγα μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω τις δικές μας τις τροπολογίες και των σοσιαλδημοκρατών να τις στηρίξετε. Ευχαριστώ. Ο έχει το λόγο εκ μέρους ε, της Ευρώπης Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό των προϊόντων ε, διπλής χρήσης ε, επανέρχεται πολύ συχνά στη συζήτηση. Είναι σημαντικό γιατί για να εξαχθεί οποιοδήποτε προϊόν στον κατάλογο το προϊόντα διπλής χρήσεως στη Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται να λάβει πρώτα άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιολογεί αυτή την προϋπόθεση με το επιχείρημα ότι ο κατάλογος των προϊόντων διπλής χρήσης ε, αποτρέπει την ε, δρομολόγηση όπλων που μπορούν να καταλήξουν σε χέρια δικτατόρων. Θυμάστε όμως τι έγινε με τον Καντάφη. Εκεί είχαμε ε, όπλα 320 εκατομμύρια ευρώ που έφτασε στα χέρια του μέσα σε μία πενταετία. Οπότε το επιχείρημα που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αφενός αβάσιμο και άστοχο και αφετέρου και υποκριτικό. Για να είμαστε λοιπόν σαφείς, στόχος της πρότασης αυτής είναι να εκχωρήσει ακόμη μεγαλύτερες εξουσίες και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αποφασίζει ποια προϊόντα θα ενταχθούν στον κατάλογο των προϊόντων διπλής χρήσης. Η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα έθνος που υποστηρίζει το παγκόσμιο εμπόριο. Λοιπόν, θεωρώ παράδεκτο μη εκλεγμένοι γραφειοκράτε να ε, ρυθμίζουν ε, τις εξαγωγέ του Ηνωμένου Βασιλείου και μάλιστα να απαγορεύουν μερικές φορές και τις εξαγωγέ συγκεκριμένων προϊόντων. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο ε, Σούστα. Αλλά... Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να πάρω ένα λεπτό από, την, ε, τον χρόνο του κύριου Σούστα. Ο κύριος Σούστα δεν μπορούσε να έρθει και νομίζω ότι μπορώ να ήταν, θα ήταν σύμφωνος να μου δώσει αυτό το χρόνο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Catch θα έχετε το ένα λεπτό αυτό το οποίο ζητάτε. Αλλά τώρα ο κύριος, ε, ο κύριος Τσούτας έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο έλεγχο εξαγωγών για προϊόντα διτή χρήση είναι απαραίτητο ώστε να αποτρέψουμε την ε, διασπορά ε, οπλικών συστημάτων. Και φυσικά είναι και εμπορικό το συμφέρον γιατί είναι, τα, είναι προϊόντα τα οποία μπορούν να τύχουν εμπορίας για πολιτικού στόχου, για μη στρατιωτικού στόχους. Γι' αυτό χαιρετίζουμε την ε, πρόταση της Κομισιόν και είναι καιρός πια να υπάρξει η σωστή εφαρμογή αυτών των μέτρων. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα προϊόντα και αυτές τις τεχνολογίες θα εξάγονται με τρόπο ο οποίος δεν θα παραβιάσει θεμελιώδεις ελευθερίες και τα θεμελιώδη <clears throat> δικαιώματα και επομένως η παροχή τεχνολογιών που αναφέρονται σε εφή τηλέφωνα κτλ. δεν θα μεταλαμβαδεύεται με τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Και τελευταίος ο κύριος Λάιχτφριντ έχει το λόγο και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να αναφέρω, ε, να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ελέγχθη προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι αληθεύει. Για τον κανονισμό αυτό για τα προϊόντα διτής χρήσης δεν πρόκειται να εμποδίσουμε τις εξαγωγές από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς θέλουμε να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εξαγωγείς. Και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι διαφορετικό από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Είναι μια χώρα η οποία έχει τους δικούς του κανόνες οι οποίοι είναι απόλυτα συνεπείς αλλά δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως ισχύουν στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει ο είναι να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο καταρχήν όλοι συμφωνούμε. Και υπάρχουν και πλεονεκτήματα τα οποία θα προσποριστεί η Μεγάλη Βρετανία από το εμπόριο αυτό στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δημιουργεί λοιπόν μια ευκαιρία και για το Ηνωμένο ο κανονισμός. Ευχαριστώ κύριος Όμπερ Μάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα προϊόντα αυτά διπλής χρήσης είναι τεχνολογία και αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολιτικούς και στρατιωτικούς λόγους όπως υπολογιστές και ε, αντικείμενα διαστημικής. Οποτεδήποτε γίνεται αυτό θα πρέπει να το εμποδίζουμε κυρίως στη στρατιωτική χρήση. Από την άλλη όμως πρέπει να μην περιορίσουμε υπερβολικά το νόμιμο εμπόριο. Επειδή λοιπόν τα τεχνολογικά προϊόντα σήμερα εξελίσσονται με ταχύτητα είναι σημαντικό να έχουμε μια ταχεία και ευέλικτη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, τρίτες χώρες αντιδρούν γρήγορα και δεν πρέπει να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κατόπιν τούτου πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή, αλλά αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες πλαίσιο. Καταρχήν εξαρτάται από την επικοινωνία των αρχών των κρατών μελών μεταξύ τους, από τη συνεργασία ανάμεσα στις ελεγχόμενες υπηρεσίες και τρίτον επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογή εφαρμογής των διατάξεων. Ο Επίτροπος Δεχόχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός αυτή τη φορά. Θα ήθελα να καθησυχάσω και να διαβεβαιώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να παράσχει όλες τις σχετικές και απαραίτητες πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ετοιμάζει κατεξουσιοδότηση πράξης προκειμένου να εξασφαλίσει ε, εξονυχιστικό έλεγχο των ε, καταξιδιών της πράξεων με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Σχάκε για το λογισμικό και άλλες τεχνολογίες, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αποφύγει, να εμποδίσει εξαγωγή τεχνολογιών για παρεμβολή στις τηλεπικοινωνίες και μάλιστα υιοθέτησε και κυρώσεις κατά της Συρίας και του Ιράν. Και σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή, κύριε Πρόεδρε, μας ενδιαφέρει η ταχύτητα, ταχύτητα και αφαίρεσης ενός προϊόντος από το κατάλογο, αλλά και ταχύτητα στη συμπερίληψη ενός προϊόντος ε, στον κατάλογο αυτό της διπλής χρήσης. Και αυτό και ζητήσαμε την συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Και ο εισηγητής μας, ο κύριος Κέλνερ, θα έχει και τον τελικό λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν, δεν διαφωνούμε ως προς τα ουσιώδη ζητήματα. Κάποια προϊόντα διπλή χρήση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την καταπίεση των ανθρώπων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικού λόγου για τον πόλεμο. Γι' αυτό θα έπρεπε να συνοδεύονται από την αυστηρότερη δυνατή νομοθεσία για τον έλεγχό του. Το θέμα είναι δεν υπάρχει πια κάτι τέτοιο, γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν τροποποιηθεί οι διαδικασίες για την τροποποίηση των ε, καταλόγων αυτών και γίνονται πολύ χρονοβόρες ε, και επαχθεί. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη νέα νομοθετική πρόταση για να επισπεύσουμε τη διαδικασία και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ε, εξελίξεις. Και έτσι να αποφύγουμε την αλλαγή του συνόλου της νομοθεσία. Αυτό έχει ήδη προγραμματιστεί για αργότερα. Αλλά τώρα θα πρέπει να ενημερώσουμε το συγκεκριμένο νομοθέτημα με βάση την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε πράγμα στο καιρό του λοιπόν και ο καιρό ε, τώρα είναι να εγκρίνουμε το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, όχι να προδικάσουμε, να προεξοφλήσουμε μελλοντικέ συζητήσει. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή μα για το έργο του. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για το θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε, δεν προλάβαμε να δώσουμε το λόγο σε όλους όσους τον ζήτησαν έχουμε πίεση χρόνου γιατί στις 6 θα πρέπει να συνεχίσουμε τη διαδικασία των ψηφοφοριών.